Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ανταλλαγή απόψεων ε, με τα μέλη της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Από την ε, δημιουργία της η Επιτροπή ΔΕΒΕ ασχολείται με την πλατφόρμα για τους ε, καταναλωτές και τη θεωρεί σημαντικό κομμάτι για την προώθηση των, των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα είμαστε εδώ για να ακούσουμε περισσότερα για τη δουλειά της πλατφόρμας και, και την έκθεση που επίκειται και που θα υιοθετηθεί τον Οκτώβριο. Με 17 7 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που καλύπτουν όλα τα θέματα που αντιμετωπίζει η ανθρώπινη κοινωνία, οι χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά προσπαθούν να ε, επιταχύνουν την ε, επίτευξη πιο ε, συμπεριληπτικών προγραμμάτων μέχρι το 2030. Η Επιτροπή ΔΕΒΕ προσπαθεί να κατανοήσει την προσέγγιση του Πρόεδρου Γιούνκερ για την ε, βιωσιμότητα και το πώ προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει του στόχου τη χιλιετία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε λοιπόν πότε θα υποβάλει η Κομισιόν το σχέδιο ε, στοχασμού και να δούμε την ε, ε, ανακοίνωσή της ε, για το 2030 και την αποτελέσματα για την Συμφωνία του Περιουσιού. Οι στόχοι πρέπει να εφαρμοστούν σε παγκόσμιο επίπεδο και να παρακολουθούνται. Η υποβολή εκθέσεων επίσης για το 2019 και το σχετικό πολιτικό φόρουμ υψηλού επίπεδου είναι άλλο ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο θα θέλαμε να αναφερθεί η Κομισιόν και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μακάβων, πρόεδρο της Επιτροπής ΔΕΒΕ, η προσκεκλημένη μας. Καλώς ήρθατε και αναλάβετε τα ενία. Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Βαλάν, που μας, καλέσατε στη σημερινή συνεδρίαση. Η Επιτροπή μας ε, εμπλέκεται στου στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, παρακολουθεί τις ε, συναντήσεις υψηλού επίπεδου στη Νέα Υόρκη ήδη από το 2015 και του Πολιτικού Φόρουμ, από τότε δηλαδή που υιοθετήθηκαν οι ε, στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης. Βρισκόμαστε στην τρίτη τους επέτειο, είναι τριών χρονών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση α, ήθελε να πιέσει για την, στη Νέα Υόρκη για την επίτευξη των στόχων αυτών και το πιο σημαντικό για τη δική μας Επιτροπή είναι ότι ναι, δουλεύουμε τις εξωτερικές πτυχές της εφαρμογής των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και το κάνουμε έτσι ώστε να έχουμε ε, συμφωνία για, τα, για την ανάπτυξη για άλλα εργαλεία, αλλά και για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα τελικά συνολικά για τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Γιατί σε πολλά υπουργεία σήμερα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες, οι πολίτες θεωρούν τους στόχους ως υποκατάστατο των στόχων της χιλιετίας και το, σκεπτικό των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης είναι, ένας, ε, είναι ο κοινό μας πλανήτης με τους κοινού πόρους και πρέπει να δούμε όλες τις πολιτικές σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλες τις χώρες. Είναι λοιπόν αλλαγή νοοτροπίας κυρίως για τη βιωσιμότητα και ελπίζω ότι σήμερα θα Έχουμε κάποιες ε, πληροφορίες από τους εμπειρογνώμονές μας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το πώς, γιν, πώς ξεκινούν οι ε, προετοιμασίες για τον Ιούλιο του 2019, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει την έκθεσή της για το πώς η ίδια εφαρμόζει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και ε, επίσης θα ήθελα να ακούσουμε τι γίνεται με τι εξωτερικέ αλλά και με τι εσωτερικέ πτυχές και πώ αυτέ θα καταγραφούν στη Νέα Υόρκη. Γιατί το Κοινοβούλιο δεν είναι πολύ εύκολο αυτό το χρονικό σημείο γιατί είναι και οι ευρωεκλογέ την επόμενη Μάιο, θα έχουμε νέο ε, Κοινοβούλιο αρχέ του Ιουλίου, οπότε είναι λίγο σαφέ ακόμα πώ θα γίνει, πώ θα λειτουργήσει όλο αυτό, Κυρίω ό,τι αφορά την εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου. Οπότε το 2019 και το 2018 ότι παραμένει, αλλά και το επόμενό έτος πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως Κοινοβούλιο για να πιέσουμε ώστε να υπάρξει σωστή προετοιμασία για αυτή την εκδήλωση. Την επόμενη εβδομάδα υπάρχει μια αντιπροσωπεία που θα πάει στη Νέα Υόρκη. κάποια από τα μέλη της είναι εδώ στην ε, αίθουσα και βεβαίως θα ήθελα να καλωσορίσω και τους ε, ομιλητές. Θα ακούσουμε καταρχάς τον εκπρόσωπο της πλατφόρμας ε, για, τις, για τους στόχους βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα τη Επιτροπή για να μα πει πώ ε, τα οργανώνει όλα αυτά, τι εσωτερικέ και εξωτερικέ πτυχέ η Κομισιόν. Θα ακούσουμε το, την Υπηρεσία περιβάλλοντο του ΟΗΕ και μετά την Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ και την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Ξεκινούμε λοιπόν από την πολυμερή πλατφόρμα για τους στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο κύριο Γιάν Νότερνταμ από το CSI Europe ο κύριος Κόρμπι από την Επιτροπή ε, των Περιφερειών και η κυρία Πατρίτσια Χέδιγκερ από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει πρώτος το λόγο. Και αν μπορείτε κιόλας να πείτε στην Επιτροπή τι είναι ακριβώς η πλατφόρμα, η πολυμερής πλατφόρμα, πώς λειτουργεί και πώς θεωρείτε εσείς ότι εμπλέκεστε στην όλη εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, so... Σας ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Πατρίσια Χάιντεγκερ. Θα αρχίσω εγώ. Έχουμε μια, κενή, έχουμε μια κοινή παρουσίαση για τους στόχους της ε, πολυμερούς ε, πλατφόρμας. Ξέρετε ότι η πολυμερής ε, πλατφόρμα ορίστηκε από την πρώτη συνάντηση πέρσι το Δεκέμβριο η πλατφόρμα αυτή είναι μία πλατφόρμα ε, που απαρτίζεται από εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες. Υπάρχει ε, το μέρος των ανώτατων αξιωματούχων, δηλαδή του υψηλού επίπεδου και εμείς που αναλαμβάνουμε την καθημερινή εργασία. Ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που μας απασχολεί. Αυτή τη στιγμή μας απασχολεί ένα συγκεκριμένο θέμα, όχι και μοναδικό, δηλαδή το πόσο έχει συνεισφέρει η πολυμερής πλατφόρμα στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο έγγραφο συλλογής. Και θα συντάξουμε αυτό το έγγραφο σκέψεων και περισυλλογής και θα σας δώσουμε τα τελικά συμπεράσματα που θα είναι έτοιμα τον Οκτώβριο. Θα σας πούμε πού βρισκόμαστε μέχρι ε, τώρα. Έχουμε έξι υπόμαδες, άρα είναι μια συνεχής διαδικασία πέρα από το έγγραφο περισυλλογής. Για το επόμενο πολιετές θα υπάρξει ένα έγγραφο για τη βιωσιμότητά του και πώς θα επιτευχθεί και θα ήθελα να πω ότι η εργασία στο MSP αποτελεί πραγματικά ε, μία πολυμερή πλατφόρμα, κοινωνία των πολιτών, ε, συμβούλια και κοινότητες, τοπικές αρχές, εργοδότες, καταναλωτές αλλά υπάρχει μια πρώτη προστιθέμενη αξία, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια αίθουσα και προσπαθούν να βρουν κοινέ λύσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διαδικασία που ανοίγει πόρτες προς διάφορες κατευθύνσεις για να μάθουμε ημένα από τους δε και να βρούμε λύσεις. Λοιπόν, τώρα θα σας παρουσιάσω την εργασία μας όπως σας είπα, είναι προκαταρκτικές οι συστάσεις γιατί η πολυμερής πλατφόρμα μόνο τον Οκτώβριο θα αποφανθεί επί του εγγράφου περισυλλογής της Επιτροπής, άρα σας μιλάμε για αυτή την εργασία που εξελίσσεται. Έχουμε πέντε κεφάλαια και θα σας τα παρουσιάσουμε εντάχει και οι τρεις Θα αρχίσω με το πρώτο κεφάλαιο που είναι το όραμά μας. Πριν φτάσω σε ένα από τα σημεία ε, κλειδιά, δηλαδή η, μια βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030, θα ήθελα να τονίσω ότι από τη μία πλευρά Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την Ατζέντα 2030 και τους βιώσιμους ε, στόχους ανάπτυξης και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο για να έχουμε ένα θετικό αφήγημα για την κοινωνία μας, έτσι ώστε όλοι να κατανοούν το επίγον της ε, άμεσης δράσης, τον επίγοντα αυτό χαρακτήρα και προσπαθούμε να θέσουμε ευρωπαϊκά πλαίσια βράσης για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μέσα στα πλαίσια ε, του NDG+. Και γι' αυτό προσπαθούμε να δούμε τι σημαίνουν οι συγκεκριμένοι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μπω σε όλα τα στοιχεία Μπορείτε να διαβάσετε και την έκθεσή μας όταν είναι έτοιμη. Όμως υπήρχε συνένεση ότι θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις και ποια θα είναι η ιεράρχησή μας των στόχων. Επίσης, έχουμε ορίσει ορισμένες βασικές αρχές μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών δεδομένων. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν πίσω. Αυτή είναι η βασική αρχή. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για την εξωτερική δράση και την ε, συνεργασία, την αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά μας ενδιαφέρει και στα πλαίσια των εσωτερικών πολιτικών. Ένας άλλος βασικός στόχος είναι η συνδεσιμότητα των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλές φορές δεν υπάρχει συνδεσιμότητα, άμεση συνδεσιμότητα. Δηλαδή το κίνημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν, συμμέχει, δεν συμμετέχει δραστικά στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Πώς μπορούμε να κάνουμε λοιπόν αυτή τη συνδεσιμότητα. Μια άλλη βασική αρχή είναι η συνοχή για την αναπτυξιακή πορεία μας. Θα επανέλθουν οι συνάδελφοι επί του θέματος, όμως υπάρχει μεγάλη πρόκληση για μας για να υπάρχει μία ενιαία πολιτική για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι ότι χρειαζόμαστε μία στρατηγική για την Ευρώπη του 2030, άρα υπάρχει ευρεία συνένεση στην πολυμερή πλατφόρμα για να έχουμε μία στρατηγική που εποπτεύει τα πάντα και υπάρχουν ορισμένα άλλα βασικά στοιχεία θα πρέπει να, είναι, να έχει ένα όραμα και να ε, είναι μετασχηματιστή και να μας δώσει έναν οδικό ε, χάρτη με συγκεκριμένους στόχους μέχρι το 2030 να καλύπτει τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές. Θα πρέπει να βασίζεται σε μία εις βάθος ανάλυση για τα χάσματα που υπάρχουν λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να κινείται πέρα από το πενταετές πλαίσιο να είναι μακροπρόθεσμη στρατηγική, να ε, δει τη συνδεσιμότητα μεταξύ βιώσιμων στόχων, να μην είναι επιλεκτική η πολιτική, να καλύπτει και τους ε, τέσσερους, ε, τέσσερις τομείς, τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό και τις διαστάσεις διακυβέρνησης. Επίσης θα πρέπει να εποπτεύει ποιοτικά και ποσοτικά την πρόοδο προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, θα πρέπει να μετασχηματίσει τα οικονομικά και κοινωνικά πρότυπα, καθώς και να προβάλλει ένα ε, υπόδειγμα μετασχηματισμού. Και τέλος, θα θέλαμε, θα θέλαμε να, γίνουν, να γίνει μια αξιολόγηση της πολυμερούς πλατφόρμας και να δούμε κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει ένα πάγιο μέσο για να παρακολουθήσει τη διαδικασία μέχρι το 2030. Θα δώσω τώρα το λόγο στο συνάδελφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πατρίτσια. Και για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η στρατηγική, βιώσιμη στρατηγική για την Ευρώπη του 2030, δεν θα καταφέρουμε τίποτα χωρίς πιο ισχυρή ηγεσία και χωρίς αναθεώρηση της ε, διακυβέρνησή μας. Ε, να επαναλάβω δύο πράγματα που περιλαμβάνονται εδώ πέρα στην έκθεση για τις προσδοκίες προς την ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την Επιτροπή προτείνουμε στην Επιτροπή να υπάρχει μία ομάδα ειδική και ο πρόεδρος να είναι υπεύθυνο για την σωμάτωση των ε, στόχων της χιλιετίας, των στόχων των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων σε όλες τις άλλες πολιτικές. Αυτό προφανώς θα σημαίνει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και να πούμε ότι η εμπειρία κάποιων υποομάδων που εργάζονται στην πλατφόρμα καταδεικνύει πολύ θετικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την σχέση μεταξύ των υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά παρατηρούμε ότι αυτό ισχύει και σε διάφορες υπηρεσίες. Υπάρχει μεγάλη όρεξη προκειμένου να πετύχουμε μεγαλύτερη συνέχεια, συνοχή και αντίκτυπο. Πιστεύουμε ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να αξιολογεί την πρόοδο που σημειώνεται και να διαγράφει τις περαιτέρω που χρειάζονται σε ό,τι αφορά τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους στην ετήσια έκθεση ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης που εκφωνεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης να αναφέρει τα σχετικά στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Αυτή είναι μια προσδοκία εντονότατη την οποία προβάλλουμε. Δεν γίνεται να υπάρχει έκθεση για την κατάσταση της Ένωση χωρίς δήλωση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τα επόμενα βήματα σε αυτό το σημαντικό στοιχείο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, Κοινοβούλιο, συγγνώμη, συνομοθετή. Φαίνεται ότι είναι και μια λογική, αλλά υπάρχει μεγάλη προσδοκία προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει ότι οι βιώσιμοι δεξιακοί στόχοι ενσωματώνονται με ομογενή, ομογενή τρόπο σε όλα τα ζητήματα, σε όλου του φακέλου όλων των επιτροπών. Πώ θα οργανωθείτε λοιπόν στο Κοινοβούλιο, με ένα πιο εγκάρσιο τρόπο σε όλες τις επιτροπές, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις αυτό θα αποτελούσε μεγάλη πρόκληση. Το ίδιο συμβαίνει και στις κυβερνήσει, στις μεγάλες επιχειρήσεις, στην Επιτροπή. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν συνοχή και ομοιογένεια στο έργο των διαφόρων ομάδων και επιτροπών. Επίσης υπάρχει μια προσδοκία και η εμπλεκόμενοι φορεί υπολογίζουν στους βουλευτές προκειμένου να διαπαιδαγωγήσουν και το εκλογικό τους κοινό και τη, να υποστηρίξουν και την, τον εντοπισμό των βιώσιμων στόχων. Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινή ζωή των πολιτών, των επιχειρήσεων και άλλων ε, βασικών φορέων στην κοινωνία. Επίσης υπολογίζουμε να υπάρξει ένα ισχυρή από το Κοινοβούλιο προς την Επιτροπή για να δοθεί κίνητρα χρηματοδότησης για την ανταλλαγή καλών πρακτικών για να ενθαρρυνθούν και οι δήμοι, οι κοινότητες, οι περιφέρειες και τρίτες χώρες για να εφαρμόσουν τους ε, βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους αυτά και να καλέσω τον Μπέρτ να πάρει το λόγο σε ό,τι αφορά το τρίτο κεφάλαιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάω το τρίτο κεφάλαιο. Εδώ κοιτάμε πώς χρησιμοποιούμε το, την εργαλειοθήκη σε πέντε βήματα. Καταρχάς, ένα βασικό στοιχείο είναι ο ορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και εδώ έχουμε την αίσθηση ότι είναι απαραίτητο η βιώσιμη ανάπτυξη να είναι στο επίκεντρο των μελλοντικών πολιτικών και των πολιτικών κατευθυντηρίων γραμμών όλων των θεσμικών οργάνων. Πενταετής περίοδος ε, κατευθυντήριων γραμμών σε ό,τι αφορά τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Και με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε και κάποιες ιδιαίτερες ε, προκλήσεις, όπως είναι για παράδειγμα η Ατζέντα 2030, η η στόχη, μέσω ομοιογένειας της πολιτικής. Μόνο λοιπόν αν επικεντρωθούμε στην στη βιώσιμη ανάπτυξη θα καταφέρουμε να πετύχουμε συνοχή. Και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όλοι οι παράγοντες είναι ενήμεροι. Το θέμα λοιπόν είναι να υπάρξει ευαισθητοποίηση και των πολιτικών και των ε, δημοσίων υπολειλών. Στην επόμενη φάση έχουμε την κατάρτιση πολιτικής. Εδώ είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι οι βιώσιμοι στόχοι, οι βιώσιμοι στόχοι, θα ενταχθούν σε όλη τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προσαρμογή της ε, ατζέντα για την καλύτερη νομοθεσία, προκειμένου να είναι επαρκή αλλά και κυρίω συνεκτική η νομοθεσία και εδώ η συνοχή αποτελεί εκ νέου πρόκληση. Να θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό με μια υποχρέωση πρωταρχική να υπάρχει βιωσιμότητα και αυτό να μπει σε όλες τις πτυχές της νομοθετικής απόφασης. Τρίτο βήμα. Κύκλος πολιτικού συντονισμού, Θα τα δούμε και σε ξεχωριστή διαφάνεια. Αλλά το θέμα εδώ είναι να εισαχθεί μια νέα βιώσιμη Ευρώπη σε έναν κύκλο συντονισμού. Χρηματοδότηση. Και εδώ θα υπάρξει ξεχωριστή διαφάνεια. Το θέμα λοιπόν είναι να υπάρξει σωστή χρηματοδότηση και οικονομικά κίνητρα. Όχι μόνο λοιπόν οικονομική βοήθεια και χρηματοδότηση, αλλά και φορολογικά κίνητρα. Και τέλος, παρακολούθηση, λογοδοσία και αναθεώρηση για να υπάρχουν τα σταθετικά στοιχεία, οι δείκτες που χρειαζόμαστε σε ένα σύστημα το οποίο θα εξασφαλίζει τη λογοδοσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Να κοιτάξουμε λοιπόν στα γρήγορα το νέο κύκλο συντονισμού πολιτικών που προτείνουμε, που βασίζεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, σε μία γενικότερη στρατηγική για την Ευρώπη του 2030 που αποτελεί και την γενικότερη στρατηγική που μας καθοδηγεί για όλες μας τις πολιτικές. Αυτό λοιπόν θα αφορά και τον υφιστάμενο κύκλο πολιτικής όπως τον γνωρίζουμε και θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταστεί πιο βιώσιμος και ένα νέο κύκλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην δεξιά πλευρά τα δύο στοιχεία αυτά λοιπόν είναι ενσωματωμένα και με μία ετήσια έρευνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα καθορίσει και τις προτεραιότητες και σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε μια εθνική ε, διαδικασία κατάρτισης σχετικών εξαίσεων και στα αριστερά βλέπετε σε ένα κύκλο τετραετή-πενταετή που θα τροφοδοτεί και το εξάμεινο το οποίο θα καταστεί πιο βιώσιμο μιας και θα υπάρχει και ένας έλεγχος βιωσιμότητας. Χρηματοδότηση τώρα και παρακολούθηση. Εδώ το σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο θα δραματίσει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την βιώσιμη διαμόρφωση της χρηματοδότησης και από την δημοσιονομική πλευρά, αν και αυτό αποτελεί πιο πολύ καθήκον των κρατών μελών και σε ό,τι αφορά τις πιο βιώσιμες δημόσιες δαπάνες, προκειμένου να υπάρξει επικέντρωση και στον ιδιωτικό τομέα και στην ιδιωτική χρηματοδότηση σε πιο βιώσιμες πρακτικές. Συνομοθέτης λοιπόν και κοινοβουλευτικός ελεγκτής. Και στα αριστερά βλέπετε, στα δεξιά μάλλον του γραφήματος βλέπετε το σύστημα παρακολούθησης το οποίο θα πρέπει να ισχύει σε όλες τις πολιτικές, σε όλες τις επιτροπές, όχι μόνο με ποσοτική αλλά και ποιοτική ανάλυση. Αυτό ας το προσπεράσουμε, μιας και το είδαμε σε προηγούμενη διαφάνεια και να δώσω το λόγο πάλι σε εσά. Η παρέμβασή μας έχει και ένα κομμάτι που φορά στις συγκεκριμένες ε, πολιτικές προτάσεις. Ε, έχουμε τα θέματα των αδομών της διαχείρισης, έχουμε το ευρωπαϊκό, την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, αλλά είδαμε ότι ε, ήταν, είναι σημαντικό να γίνουν πιο συγκεκριμένα τα πράγματα και να δείξουμε τι ακριβώς ε, σημαίνει η πολιτική προσέγγιση στο πρόγραμμα λοιπόν αυτό για τις προτάσεις της ε, πολιτικής θέλαμε να τονίσουμε ότι η βιωσιμότητα θα πρέπει να, να αντικατοπτρίζεται με συνεκτικό τρόπο σε όλη την ευρωπαϊκή ατζέντα αναφέροντας και τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και τις διάφορες προοπτικές οπότε οι προτάσεις που, που κάνουμε δεν είναι ε, διεξοδικές ε, προσπαθούμε να βρούμε κάποιες ομάδες προτάσεων. Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να ε, μελετούμε ανά τομέα πολιτικής τις προτάσεις, αλλά να υπάρξουν κάποιες ομάδες ανά πρόκληση που έχουμε καταγράψει. Αυτά είναι ε, απλώς ε, παραδείγματα που σας δείχνω εδώ. Ε, υπάρχουν προσεγγίσεις από τα κράτη-μέλη για τις, τις δικές τους εκθέσεις, όπου καθορίζουν κάποιες συγκεκριμένε ομάδες πολιτικής, τομείς δηλαδή, και δείχνουν πώς μπορούν να υπάρξουν, να καλυφθούν πιο συνεκτικά τα θέματα τα, κλιματοικά, του περιβάλλοντος κτλ. Θα σας δώσω εγώ τις δικές μας προτάσεις για τους πέντε τομείς που έχουμε καταγράψει, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πολιτική με διάφορα παραδείγματα. Υπάρχει λοιπόν ένας τομέας που αφορά στην βιώσιμη παραγωγή και την κατανάλωση, που σημαίνει κυκλική οικονομία, αλλά όχι μόνο, Έχουμε μία ομάδα που αφορά στην ε, κοινότητα και την ε, ε, συμμετοχή, επίσης απασχολησιμότητα και κοινωνική ενσωμάτωση, ένταξη. Έχουμε την ομάδα που ασχολείται με την ενέργεια και το κλίμα προφανώς και πάλι εδώ συνδεόμαστε με άλλους τομείς πολιτικής που έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο. Τέταρτο, τρόφιμα, παραγωγή, ε, χρήση και γεωργία. Δεν περιοριζόμαστε μόνο στην ΚΑΠ, αλλά γενικώ μιλούμε για το, συνολικά για το πρόγραμμα ε, παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων. Και τέλος, πολιτική συνοχής. Αυτοί είναι οι πέντε βασικοί τομείς τους οποίους έχουμε καταγράψει και δίνουμε κάποια παραδείγματα συστάσεων πολιτικής που δείχνουν πώς θα μπορούσαμε να τα δούμε πιο ολοκληρωμένα όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν θα μπω σε άλλες λεπτομέρειες. Απλώς ήθελα έτσι να σας δείξω μια γενική εικόνα της μεθοδολογίας που ακολουθούμε. Ευχαριστώ. Για το κεφάλαιο 5... εδώ να ξεκινήσω με αυτό που είπε η Πατρίτσια στην αρχή. Μετά από έξι μήνες εντατικής δουλειάς, καταφέραμε να καταλήξουμε ε, σε έναν οδηγό 260 σελίδων. Αν έχετε χρόνο το, στις διακοπές σας, διαβάστε τον, με τη συμμετοχή διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων από τα κράτη-μέλη, ε, όπου αναφέρονται οι επιλογές που έχουμε, οι συστάσεις, οι προσδοκίες. Είναι πραγματικά εμβριθές το κείμενο και ελπίζω ότι είμαστε ε, θα ήθελα μάλλον να είμαστε όλοι στις, στην ίδια, στο να έχουμε το ίδιο σκεπτικό, αλλά ε, υπάρχουν και αποκλίνουσε απόψει, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω, πρέπει να τα διαπραγματευτούμε λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό που είναι σαφέ είναι ότι αυτό που τελικά καταφέραμε να έχουμε δείχνει ότι πέραν των εντάσσεων που μπορεί ακόμη να υπάρχουν, η δέσμευση να κινηθούμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση είναι πολύ πιο ισχυρή. Και θεωρούμε ότι έχουμε πραγματικά προστιθέμενη αξία και ο ρόλος μας είναι σημαντικός και θα συνεχίσει να είναι σημαντικός και πέραν του 2019 για να εξασφαλίσουμε ότι ο πλούτος αυτός της εμπειρογνωμοσύνης και της ε, επιτόπου ε, εμπειρία μπορεί να τροφοδοτήσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και επίσης σε αυτή την πολύ δύσκολη δουλειά θα βοηθήσει ώστε να υπάρξει περισσότερη συνεκτικότητα στην πολιτική ώστε να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο. Επίσης μπορέσαμε να εργαστούμε πολύ στενά με τη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως για, την, για τη δημιουργία του προγράμματος για, την, για το ε, βραβείο βιωσιμότητας διαφόρων κατηγοριών. Υπάρχουν ε, οι προθεσμίες για την, για την κοινωνία των πολιτών και και άλλες κατηγορίες ε, μέχρι το Σεπτέμβριο και το πρώτο βραβείο θα δοθεί νομίζω τον, το, την άνοιξη του 2019. Ε, τα μέλη λοιπόν των θεσμικών, οργανώ, θεσμικών οργάνων, τα μέλη της πλατφόρμας, η κοινωνία των πολιτών θα έχουν την ευκαιρία να εκτιμήσουν τη δουλειά που έκαναν οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν εντατικά από όλες τις τοπικές κοινότητες και κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είναι αυτοί που δρούν πραγματικά και που μεταφράζουν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης σε ε, απτές λύσεις. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι οι στόχοι δεν θα γίνουν ε, ένα στοιχείο που θα παραγωνιστεί και θα αφορά μόνο στις Βρυξέλλες ή στη Νέα Υόρκη ή αλλού, αλλά έχει, είναι κάτι που μας αφορά όλους και πραγματικά τα καταφέραμε με αίμα και υδρότα να το πετύχουμε. τέλος, υποβάλλουμε την πρόταση να συνεχιστεί η προσπάθεια, να συνεχιστεί η δουλειά της πλατφόρμας, για τους λόγους που σας ανέφερα. Κάτι που δεν έχουμε καθόλου χρόνο να το συζητήσουμε και που ήταν σαφής η ερώτηση που έθεσε ο κύριος Τίμερμαν στην, εντολή, Τίμερμαν στην εντολή που έδωσε στα μέλη της πλατφόρμας είναι ποια είναι τα μέτρα που προτείνουν οι εμπλεκόμενοι φορείς ώστε οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης και όλη η διαδικασία να γίνει πιο συμμετοχική και να συμπεριλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Εδώ θα πρότεινα να πάμε πίσω στις προτάσεις που έχουν υπάρξει και έχουν ενοποιηθεί σε αυτό τον ε, οδηγό που σας ανέφερα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε μετά τη συνάντηση του Οκτωβρίου της πλατφόρμας και ίσως και αργότερα το 2019. Αλλά αυτό είναι το ερώτημα κλειδί. τι σημαίνουν αυτοί οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης για τους πολίτες. Αν σημαίνουν κάτι για τους καταναλωτές, για τους άντρες και τις γυναίκες που δουλεύουν στις δημόσιες υπηρεσίες ή στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί ούτως ή άλλως το εγχείρημα είναι κοινό για όλους. Υπάρχει μια πρόταση για να υπάρξει το ευρωπαϊκό έτος των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, είτε το 2022 είτε το 2027. Um, Βέβαια, το θέμα είναι πώς μπορούμε να συνδέσουμε τα επόμενα 65 ή 70 χρόνια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος με ένα μήνυμα κλειδί, ότι η βιωσιμότητα είναι ο θεμέλιος λίθος για τη μελλοντική ειρήνη, ευημερία και ηγεσία στον κόσμο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Well, been working for a short time, but clearly been um, busy and have some very ναι, ελπίζω να έχετε συγκεκριμένες προτάσεις σε καιρό. Είμαι σίγουρη ότι οι βουλευτές ε, θα έχουν πολλές ερωτήσεις. Ο κύριος Μαρσέλ Χάγκ είναι ο επόμενος ομιλητής από, την, ε, από πλευράς Επιτροπής, ε, του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής ε, καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε συντονισμό και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς αυτό το έγγραφο περί ε, θα μας δώσει απτά στοιχεία. Στο, στη διάσκεψη στο Συμπίου θα το θίξουμε αυτό το ζήτημα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να λάβω το λόγο. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι προσδεδεμένη στις συνθήκες της Ευρώπης και βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε η εμπροστοφυλακή της βιώσιμης ανάπτυξης και η Επιτροπή θα ήθελε να ισχύσει αυτό και στο μέλλον και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει στον ηγετικό ρόλο βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Επιτροπή αυτή εργάζεται για την εφαρμογή της Ατζέντα 2030 σε επτά τομείς. Ο πρώτος ορίστηκε στην ανακοίνωση του Νοεμβρίου του 2016 που έχει ήδη υποβληθεί και συζητηθεί στο φόρουμ αυτό. Σε αυτή την ανακοίνωση η Επιτροπή προβάλλει τη στρατηγική της προσέγγιση που αφορά ε, το mainstreaming του, της βιώσιμης ανάπτυξης ε, στα παγκόσμια δεδομένα και στα παγκόσμια φόρα. Και έχουμε την εργαλειοθήκη μας προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, η Επιτροπή ε, προέβαλε μία πρόταση για το επόμενο ε, ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ που να συμβαδίζει με την ατζέντα για το 2030. Και επίσης προβάλλουμε τις σκέψεις μας για να αναπτύξουμε ένα πιο μακροπρόθεσμο όραμα. Μετά το 2020 και η Επιτροπή το κάνει αυτό μέσω του εγγράφου περισυλλογής και σκέψης, το οποίο αναφερθήκατε ε, και στο οποίο βασίζεται και η πολυμερής πλατφόρμα. Το έγγραφο περισυλλογής θα ορίσει ένα πολιτικό όραμα έτσι ώστε να προωθήσει τη συζήτηση στα πλαίσια του μέλλοντος της Ευρώπης. Αυτό αποτελεί μέρος της ε, συλλογιστικής της Επιτροπής ε, Juncker μέχρι τις ευρωεκλογέ του Μαΐου του 2019 και πέραν αυτών και στόχος είναι να ενημερώσουμε και την επόμενη Επιτροπή στο τέλος του επόμενου έτους. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει σε αυτή την συλλογιστική και θα συνδράμει άμεσα. Το έγγραφο περί συλλογής θα εγκριθεί προς το τέλος του έτους, έτσι ώστε να έχουμε χρόνο για τις σκέψεις αυτές και τη συζήτηση που θα ενταχθεί στην όλη διαδικασία που θα οδηγήσει στις επόμενες εκλογές το Μάιο του 2019. Ακριβώς επειδή η Επιτροπή είναι πεπισμένη ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν ένα κοινό μέλημα που δεν αφορά μόνο τις δημόσιες αρχές αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς, ε, προέβαλε αυτή την πολυμερή πλατφόρμα για την προώθηση των ε, βιώσιμων στόχων ε, και πιστεύω ότι Έχουμε ε, περίπου 30 κράτη, μη κυβερνητικές, ε, κοινωνία των πολιτών, επιχειρήσεις ε, και multimedia που εκπροσωπούν το, την εργασία προς τα μέσα και προς τα έξω. Έχουμε συνδράμει όλοι σε αυτό το έγγραφο περισυλλογής όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, η τέταρτη δράση αφορά την εποπτεία και την αξιολόγηση. Μέσα στα πλαίσια αυτά η εποπτεία της Ατζέντα 2030 αποτελεί ε, ένα βασικό στοιχείο της εργασίας μας για να φτάσουμε στους ε, βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Είμαστε υπέρ μιας εύρωστης και ενημερωμένης διαδικασίας για να προσαρμόσουμε την ε, προσαρμογή μας όπως χρειάζεται. Υπό αυτή την έννοια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την εργασία της πολυμερούς πλατφόρμας καθώς και της ε, Επιτροπής Ανώτατων, Ανώτερων Αξιωματούχων. Έτσι θα έχουμε μία προοδευτική ενημέρωση με βάση ε, ενδιάμεσους απολογισμούς για την εφαρμογή εγκινήσει της Ατζέντα 2030 και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα μας δώσουν μια κοινή έκθεση για την Ευρωπαϊκή Συνένεση καθώς και τις επιπτώσεις της ε, ενόψης της Ατζέντα 2030. Αυτή θα είναι μια συνεισφορά προς το HLPF και θα συναντόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα ξεκινώντας από το 2019. Έτσι θα γίνουν συζητήσεις σε σχέση με αυτό το έγγραφο σκέψεων και περισυλλογής ε, και αυτό θα γίνει και στη Νέα Υόρκη. Επίσης από πέρσι Επιτροπή ε, συντάσσει μια ετήσια έκθεση εν ώψη του 2030 με βάση έναν ε, δίκτυ της Eurostat. Η πέμπτη δράση αφορά ε, το βραβείο βιωσιμότητας που ανέφερε και η πλατφόρμα, τα μέλη της πλατφόρμας Στην ανακοίνωση του 16 ανακοινώσαμε αυτό το γραφείο έτσι ώστε να προωθήσουμε τις, ε, τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης μέσω βραβείων. Αυτό το εγχείρημα άρχισε τον Ιούνιο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως η Επιτροπή θα επιθυμούσε ε, συγκεκριμένοι και όλοι οι ευρωβουλευτές να αναφερθούν σε αυτό το βραβείο στις εκλογικές τους περιφέρειες. Ως προς τις κλιματικές αλλαγές Έχουμε την ε, νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αντιμετώπιση των καυσαερίων θερμοκηπίου ε, μετά από το Συμβούλιο του Μαρτίου και θα παρουσιάσουμε αυτή την στρατηγική το πρώτο τρίμηνο του 19. Η Επιτροπή προτίθεται να προωθήσει αυτή την εργασία και να προβάλλει ένα έγγραφο, να συντάξει ένα έγγραφο μέχρι το Σεπτέμβριο φέτος. Η Επιτροπή κατά αυτόν τον τρόπο θα ήθελε να αποστείλει ένα μήνυμα στην COP24 στην Κατοβίτσε ότι θα συνδράμουμε άμεσα έτσι θα αναζητήσουμε συνέργειες με άλλες πολιτικές και πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα την Ατζέντα 2030 και τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Η Συμφωνία των Παρισίων και η Ατζέντα του 2030 συνδέονται άμεσα. Το επικείμενο έγγραφο συλλογής για μια μακροχρόνια στρατηγική για την αντιμετώπιση των εκπομπών θερμοκηπίου θα συνδράμει άμεσα προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, συνεργαζόμαστε ως προς την εξωτερική διάσταση. Θα συνεχίσουμε να κατέχουμε ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και θα προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καταπολέμηση των ε, κλιματικών αλλαγών. Η ΚΕΠΑ ορίζει τη στρατηγική κατεύθυνση και ορίζουμε και τη συνδεσιμότητα με την Ατζέντα 2030. Τον Ιούνιο του 2017 φτάσαμε σε μια νέα συνένεση σε αυτό το επίπεδο, στο ε, φόρουμ υψηλού επίπεδου. Θα δείξουμε ότι έχουμε δεσμευτεί σε αυτή την ατζέντα εν ώψη του 2030, προβάλλοντας ε, δράσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο. η Επίτροποι Βέλα και Μίμητσα, καθώς και αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών και του ESC, θα αναλάβουν ε, ρόλο πρέσβεων. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι ότι μετά την έγκριση της Ατζέντα 2030 υπάρχει, έχει δοθεί μια μεγάλη όθηση που παραμένει. Η κοινωνία των πολιτών, οι επιχειρήσεις και οργανώσεις εστιάζουν την προσοχή στις ε, βιώσιμες ε, πολιτικές και φυσικά χρειάζεται και περαιτέρω δράση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους στόχους στόχους, ε, τους αναπτυξιακούς στόχους αυτούς και θα πρέπει να κινηθούμε βέβαιως και πέρα του 2030. Θα ήθελα να εγγυηθώ ότι η Επιτροπή ε, είναι πεπισμένη ότι θα πρέπει να παραμείνει ηγετική δύναμη στον τομέα των ε, δράσεων αυτών και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και θα ήθελα να ζητήσω από το συνάδελφο τον Κασπάρ Φοντίνη από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ να σας μιλήσει για την εξωτερική διάσταση. Ναι, Αρχίζει και αγχώνομαι γιατί έχουμε κάποιους βουλευτές που περιμένουν εδώ 45 λεπτά και δεν έχουν προλάβει να κάνουν καμία ερώτηση. Γιατί και εσείς ε, θα θέλετε να πάρετε το λόγο. Μήπως να πάρετε το λόγο αν θέλετε μετά τους ε, βουλευτές, γιατί πολλοί είναι από την Επιτροπή Ανάπτυξη εδώ να μιλήσουν πρώτα οι βουλευτές και μετά Γκασπάρ θα πάρει το λόγο, γιατί ξέρω ότι κάποιοι από του βουλευτέ θέλουν να πάρουν τώρα το λόγο, γιατί μετά έχουν και άλλες συνεδριάσει επιτροπών. Ο κύριο Τιχάρη Λουκάς έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι συντομό να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε. Είμαστε παρατηρητές σε αυτή την πλατφόρμα και να σας παρουσιάσουμε κάποια γεγονότα. Αναγνωρίζουμε αυτά που συμβαίνουν. E Πιστεύουμε ότι για να συμπεριληφθούν οι βιώσιμοι μεταξιακοί στόχοι θα πρέπει να κάνουμε πολύ παραπάνω και θα πρέπει να δράσουμε πολύ πιο γρήγορα. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε πάλι το θέμα του κλίματος. Το συζητάμε κάθε μέρα και νομίζω ότι είναι σωστή αναλογία που γίνεται μεταξύ των ε, στόχων της χιλιετίας, συγγνώμη, των, ε, της συνθήκης του Παρισιού και της ατζέντα μετά από το 2030. Αυτό όμω λείπει από κάθε δημόσια συζήτηση. σε αυτά θα πρέπει να τα προσαρμοστούν. Να σα πω πώ έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την έκθεση για του βιώσιμου αναπτυξιακού στόχου και χαίρομαι που έχουμε και την αποστολή και τη ε, ΔΕΒΕ και τη ε, άλλη επιτροπή στη Νέα Υόρκη. Μα ήταν ένα μη βιώσιμο μονοπάτι. 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ε, εγκαταστάσεις υγειονομικής σε τουαλέτες, σε πασμό νερό και τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία είναι και κρίσιμα και σε επίπεδο ευρωπαϊκών ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι το στόχο υπερθμών 7, καθαρή ενέργεια, 33 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εξάρτηση από το ξύλο και κάρβουνο για να μπορέσουν να μαγειρέψουν. Και μιλάμε για το ξύλο και το κάρβουνο, το οποίο αποτελεί μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά ε, την Αφρική. Ο υπαριθμόν αντικαστοχός οι πόλεις που αποτελούν ένδειξη της φτώχειας. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλήματα. Σε όλα τις πόλεις αυξάνεται η φτώχεια των παιδιών. 3% των γεών πλέον είναι ε, πόλεις πλέον, 20% στην κατανάλωση ενέργειας και εξαρτώνται από δασικές εκτάσεις και νερό. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις. Η βιώσιμη κατανάλωση 1,7 εκατομμύρια παιδιά πλήττει ανά και μιλάμε για 35% αύξηση που προβλέπεται μέχρι το 2020 σε ό,τι αφορά για τα επίπεδα του 2015. Τρόφιμα. Ένα τρίτο όλων των τροφίμων σπαταλάται. Τα τρόφιμα που σπαταλώνται στην ε, Ευρώπη θα μπορούσαν να θρέψουν και την Αφρική και την Λατινική Αμερική. Δύο ποικιλότητα. Απόλυες, 30 ε, πλάσιες σε σχέση με προηγούμενα ποσοστά σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γερμανία και μόνο έχουμε χάσει 75% της βιοπικιλότητας. Είμαστε λοιπόν σε έναν δρόμο μη βιώσιμο. Από το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τους στόχους, τους βιώσιμους αναπτύξεις στόχους. Τι έχει πετύχει όμως σε τρία χρόνια. Όχι αρκετά. Καταρχάς, χρειάζεται ένα ορόσημο αυτό ορόσημο για να προσμετρούνται οι πρόοδοι και αυτό θα πρέπει να προωθείται και να ε, γιατί πιστεύουμε ότι θα δώσει κίνητρο παγκοσμίω. Κατά δεύτερον, είναι σημαντική η αρχή της ε, καθολικότητας. Όσοι, όλοι σας το είπατε. Χρειάζεται πολιτική δράση τώρα. Και χαίρομαι που ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει μεγάλη έμφαση στο θέμα αυτό και εμείς ε, στον ΟΙΕΡ θα το εξετάσουμε το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και την κυρία Χάουτουλα σε ό,τι αφορά και τη δικτύωση με το Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε ότι οι δράσεις αυτές είναι σημαντικές. Κατά τρίτον, θέλουμε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να αναμειχθούν και να συμμετάσχουν ε, ενεργά, γιατί πιστεύουμε ότι αυτοί οι στόχοι δίνουν μέλλον σε όλες τις γενιές και σε όλους τους ανθρώπους και θέλουμε ευχαριστούμε για την πλατφόρμα και για το έγγραφο περισυλλογή. Δεν αρκούν όμω αυτά για να επιλύσουν την κρίση σε ό,τι αφορά του αναπτυξιακού στόχου. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ενεργή οικειοποίηση και υλοποίηση των στόχων αυτών. Θέλουμε λοιπόν ηγεσία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα στοιχεία αυτά και μακάρι να τα είχατε και ε, γραπτά. Α, τα έχουμε, μάλιστα. Θα τα στείλουμε λοιπόν στους βουλευτές τα αρνητικά στοιχεία αυτά, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Να δώσω τον λόγο στην κυρία Βαλεάν τώρα να συνεχίσει και να λάβει τα ενία της Προεδρίας. Ευχαριστώ που θα μας διαθέσετε τα στοιχεία αυτά. Συνάδελφοι, ακούτε εδώ και ώρα τις παρεμβάσεις, οπότε τώρα είναι η ώρα να πείτε τις απόψεις σας. Ο κύριος Λίτς έχει το λόγο. Πρώτος, ευχαριστώ. Είμαι μέλος της ε, ομάδας των σοσιαλιστών, είμαι από τη Γερμανία και συμμετέχω μαζί με άλλους στις τελευταίες ε, συναντήσεις στη Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστώ για την πλατφόρμα αυτή. γιατί προωθεί τις ιδέες αυτές. Ευχαριστώ πολύ τον ε, κύριο Λούκας για τις ξεκάθαρες απόψεις του μας ε, είπε ποια είναι η δική του οπτική. Εγώ δεν βλέπω πάντως να επιτυγχάνουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ακούσαμε τα στοιχεία, ε, ακούσαμε κάποιους περίεργους δείκτες που δεν βασίζονται σε εξωτερικούς παράγοντες. Οι μηχανισμοί λοιπόν και το σύστημα υποβολής εκθέσεων ακόμα είναι σε εμβριακό στάδιο. Ε, είναι λοιπόν ουσιώδους σημασίας, όπως είπατε κι εσείς, να έχουμε έναν στόχο και να έχουμε και την ικανότητα να ξέρουμε πώς θα δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό σύστημα για να το πετύχουμε. Κάθε μέρα μετράει, οπότε πρέπει να αναλάβουμε δράση. Και δύο πράγματα θέλω να πω. Μία, μία ερώτηση προς την ομάδα καταρχάς για το σχέδιο στοχασμού. Ε, είπατε ότι υπάρχει πρόοδος και μα είπατε ότι το Κοινοβούλιο μέχρι τέλο του έτου μπορεί να είναι σε επαφή και να συμμετάσχει. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ να δούμε πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε αυτό, κυρίως επειδή μιλήσατε για τα περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά και τα θέματα της διακυβέρνησης, του τέσσερις πυλώνες, για να καλύψουμε περιπτώσει όπου τα μέλη των ευρωπαϊκών κρατών μελών παρουσιάζονται ε, κυρίως από την Εστονία και την ε, Δανία για την ε, λυσίδα ε, για τα κλωστοφαντουργικά. Η Κομισιόν είπε ότι δουλεύει πάνω σε αυτά, αλλά δεν κατέληξε κάπου. Οπότε έχουμε κολλήσει από κάποιες γενικές διευθύνσεις. Η Γενική Διευθυνσή Ανάπτυξης Εμπορίου, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Οπότε το ερώτημα είναι να δούμε πώς θα υπάρξουν ίσως βέλτιστες πρακτικές που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη-μέλη περισσότερα από την Γερμανία, ας πούμε, την, ε, τις που ούτως ή άλλως έχουν πρωτοβουλίες για τα κλωστοφαντουργικά. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν να μας δείξετε κάποια καλά παραδείγματα και ίσως κάποια παραδείγματα διασυνοριακής ε, συνεργασίας η ε, συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων υπήρων ή περιοχών του πλανήτη. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε, για το έτος ε, ανάπτυξης που το είχαμε το 2015. Και θα είπατε να υπάρξει άλλο ένα έτος για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, φέτος δεν τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά αλλά έχουμε την συμμετοχή των πόλεων στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, διάφορες πόλεις της Ευρώπης, ξέρω ότι η Χαϊδελβέργη συμμετέχει από τη Γερμανία. Υπάρχει λοιπόν η προσέγγιση αυτή και θέλουν μέχρι το 2025 ίσως να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να, βοηθήσουν και άλλες πόλεις να μπουν σε αυτό το γαϊτανάκι. Ε, υπάρχει προσέγγιση λοιπόν από τις ε, πόλεις η οποία θα παρουσιαστεί και στο ΚΟΠΣ και νομίζω ότι καλό θα ήταν να υπάρξει ηγετικός ρόλος από τις πόλεις. Αλλά βεβαίω ε, να υπάρξει και ένα αίτημα από το, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίσως για το έτος 2020-2021, 2022 να έχουμε το στόχο για τους, ε, να έχουμε το έτος για τους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί όντως έχουμε μείνει πολύ πίσω. Είναι νομίζω πολύ καλή ευκαιρία αυτή. Αυτά από μένα και ευχαριστώ. Thank you very much, Ms. Um, now, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τους ομιλητές. Έχω διάφορες ε, ιδέες που μου ήρθαν μετά την παρουσίαση της ε, Κομισιόν. Με την ε, πρόταση αυτή του νέου πολίτρου δημοσιονομικού πλαισίου, η Κομισιόν έχει χάσει μια πολύ σημαντική ευκαιρία να χρησιμοποιήσει το θεματολόγιο για το 2030 ως ένα πολιτικό πλαίσιο για να ελέγξει το τι γίνεται σε σχέση με τις πολιτικές και με το που πάνε τα κονδύλια. Ε, αναφερόμενοι στους ε, στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης, δεν είναι αρκετό το να τους αναφέρουμε απλώς. Το, το νέο εργαλείο που θα έχουμε ουσιαστικά προσπαθεί να πείσει για τις ευρωπαϊκές πολιτικές αντί να προωθήσει τις, ε, και να καλύψει τις ε, αναπτυξιακές ανάγκες των χωρών εταίρων. Έχουμε τους στόχους της ε, χιλιετίας, της βιώσιμης ανάπτυξης. Αν μπορέσουμε αυτούς να τους έχουμε ως πλαίσιο για να καταδείξουμε και μια κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε με το νέο πιδελταπή, θα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πιο ισχυρή παρέμβαση για να δείξουμε και την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο στόχο της επίτευξης των στόχων μέχρι το 2030. Δεν το λέω πρώτη φορά. Εγώ ανησυχώ πολύ, γιατί η ατζέντα αυτή, το θεματολόγιο εκδίθηκε το 2015, ήμασταν όλοι πολύ θετικοί για το ορόσημο, για τη χρονική στιγμή, αλλά τώρα βρισκόμαστε σε τελείω διαφορετικό κόσμο με την ε, κρίση ε, που σοβεί, με τους διάφορους μεγάλους ε, παίχτες της κακέρα που αλλάζουν τη στάση τους. Πρέπει λοιπόν και εμείς να δείξουμε το, με το παράδειγμά μας ότι δεσμευόμαστε για τους στόχους γιατί αλλιώ δεν θα υπάρξουν ούτε πόροι ούτε πολιτική βούληση για να επιτευχθούν αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουμε θέσει. Ε, χάνει λοιπόν ε, το, τη γενική εικόνα ε, τη επίτευξη των στόχων η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως σε ό,τι φορά την ε, ε, πρικοδότηση με κονδύλια για την για την επίτευξη των στόχων συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Ζητήσαμε από την αρχή να υπάρξει ένα συνεκτικό πλαίσιο, μια στρατηγική συνολική για την εφαρμογή της ατζέντα. Ακόμα δεν την έχουμε δει. Χρειάζεται περισσότερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ένα οδικό χάρτη λεπτομερής για την επίτευξη των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε ένα ε, αυστηρό ε, μηχανισμό ελέγχου με δείκτες που θα ελέγχουν όντω, θα μετρούν όντω την απόσταση από το πού βρισκόμαστε μέχρι την επίτευξη του στόχου όχι μόνο την πρόοδο που έχουμε πετύχει, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει προσεκτικά να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των πολιτικών για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και κυρίως για τις, για τις αναπτυσσόμενες χώρες και επίσης ε, τον αντίκτυπο της ε, φορολογικής μας πολιτικής. Πρέπει να έχουμε μόνιμο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει συμμετοχή και συμμετοχική και αποτελεσματική διαδικασία. Γι' αυτό χαίρομαι που ξεκινά αυτή η πλατφόρμα οι πολυμερεί για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, ελπίζοντας ότι οι ιδέες που θα προκύψουν στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν υπόψη επαρκώς. Ένα τελευταίο σημείο. Δεν θέλω να, σα σας ακούγομαι πολύ αγχωμένη, αλλά... Ε, αναφέρατε το θέμα της ε, διάσπασης ε, της γενικής ε, εικόνας. Πρέπει να γίνει και από την πλευρά της Κομισιόν και από την πλευρά του Κοινοβουλίου πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όλοι είμαστε πολύ ευαίσθητοι για τα θέματα αυτά και η Πρόεδρος επίσης. Και πραγματικά έχουμε κάποιους μήνες ακόμα μπροστά μας και μπορούμε να δείξουμε δημιουργικότητα για την πρωτοβουλία που θα μπορούμε να αναλάβουμε για να αυξήσουμε την, την ε, ευαισθητοποίηση μεταξύ των συναδέλφων και από τις άλλες επιτροπές που μπορεί να, έχουν, να νιώθουν μια τέτοια ευθύνη και να θέλουν να παίξουν ρόλο. Ας φανταστούμε λοιπόν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, να καλέσουμε τους συναδέλφους σε συζητήσεις, να τους στείλουμε υλικό, να τους στείλουμε email, Ας εφεύρουμε λοιπόν κάτι που θα μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί για να δώσουμε το, το μήνυμα που θέλουμε πριν το τέλος της θετίας μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ενθουσιασμό σας, ο κύριος Ντάς. Σημερίζομαι την εκτίμηση της ε, Ελής. Νομίζω ότι πρόκειται για μία πολύ σημαντική πρόκληση και αυτό είναι ένα ζήτημα για να δούμε πώς μπορούμε να ε, ενσταλάξουμε το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα φόρα και τους θεσμούς. Ευχαριστώ τους ομιλητές και χαιρόμαστε ότι υπάρχει εργασία και στο τομέα της εποπτείας, καθώς και τις ε, εθνικές εισηγήσεις που παίρνουμε από τα κράτη-μέλη. Λίγα είναι τα κράτη που δεν έχουν ακόμα δώσει την εισήγησή τους, που θα δώσουν μέχρι, μέχρι του χρόνου. Αλλά είναι η πρώτη φορά που η πολυμερής πλατφόρμα συναντήθηκε με το Κοινοβούλιο εδώ αν και είχαμε την εκπροσώπησή της, εγώ ήμουνα συγητής για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης από το ε, Κοινοβούλιο και εμείς έχουμε μία έδρα στην πολυμερή πλατφόρμα. Και χαίρομαι γιατί βρισκόμαστε στην απαρχή αυτών των σχέσεων δεν θα είχε νόημα να μιλήσουμε για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης αν δεν ε, μιλούσαμε για αυτή την επίσημη ε, σχέση και συνδεσιμότητα που υπάρχει. Επίσης θέλουμε να σπάσουμε αυτό τον πενταετή κύκλο γιατί καταναλώνουμε την ενέργειά μας μέσα στα πλαίσια των θεσμικών οργάνων και του χρόνου δεν θα υπάρχει καμία αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου αυτού λόγω των εκλογών στη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν ιδέες για το πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτό τον πενταετή κύκλο και πώς μπορούμε να έχουμε εκπροσώπηση και του χρόνου από την ε, ε, από την πλευρά της πολιτικής αυτής η Eurostat BERT δεν μας δίνει στοιχεία από πλευράς ε, Επιτροπής των Περιφερειών ως προς το πολιετές θεωρώ ότι έχουμε, ε, βλέπουμε δηλαδή σαφώς ότι υπάρχει έλλειψη πολιτική, σαφούς πολιτική σε σχέση με την χρήση των ορυκτών ε, καυσίμων. Δεν προχωρούμε στο phasing out των επικινδύνων καυσίμων. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία στεγανοποίησης ισχύει πλέον, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μία οριζόντια προσέγγιση. Υπάρχουν και πολλά θετικά, αλλά έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε αν θέλουμε να φτάσουμε στους απότερους αυτούς στόχους. Η κυρία Χαουτάλα. Σας ευχαριστώ πολύ και ήταν πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία, πιστεύω. Έχει δίκιο η συνάδελφος, δεν είμαστε πάρα πολύ αριθμοί εδώ σήμερα. Από εμά όμως εξαρτάται να αποφασίσουμε πώς το Κοινοβούλιο θα προχωρήσει την ελοποίηση της ατζέντα για το 2030. Η ε, η αναπληρωματική γενική γραμματέα μα επισκέφθηκε. Ήταν τιμή μα και καταλάβαμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο. Ξέρω ότι έχετε συζητήσει του ενδεχόμενου τρόπου οργάνωση τη υλοποίηση και εφαρμογή. Αυτό που είναι σαφέ είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με την υφιστάμενη κατάσταση. Θα πρέπει να σημειώσουμε το ΜΕΣ και στο πολιτέ πλαίσιο προφανώ, το είπαν και οι δύο προηγούμενοι μιλητέ αυτό άλλωστε. Αλλά όντω πιστεύω ότι ο πιο βιώσιμος μηχανισμός από αυτούς που έχει συζητηθεί και από τους δύο προέδρους και από άλλους που έχουν επιδείξει κάποια πρωτοβουλία είναι να γίνει σύνδεση της υλοποίηση με τη δουλειά που γνωρίζουμε ήδη από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια κοινή προσπάθεια. Κανένα τομέα δεν θα εξαιρεθεί και κάποιοι θα πρέπει να λάβουν μεγάλη ευθύνη. Το πιο ρεαλιστικό μοντέλο, πιστεύω, είναι η Επιτροπή περιβάλλοντο και η Επιτροπή ανάπτυξη να συνεχίσουν να παίζουν τον συντονιστικό ρόλο που παίζουν ω τώρα. Είναι σημαντική η επίσκεψη στο υψηλό βαθμό φόρουμ την άλλη εβδομάδα γιατί εκεί θα δούμε πώς διαμορφώνονται αυτά στην πράξη. Ένα από τα σημαντικά ερωτήματα είναι το πώς θα υπάρχει συνοχή στην ιστορική και ιστορική εφαρμογή. Αυτές οι δύο πτυχές συχνά αποκλίνουν. Γίνονται κάποιες συζητήσεις ε, για μια έκθεση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Ιστορική Διάσταση υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ελπίζω να υπάρχει παρανόηση στο σημείο αυτό. Πρέπει να υπάρχει κοινή εφαρμογή και υλοποίηση εσωτερικά και εξωτερικά. Επίση, πιστεύω ότι το επόμενο φθινόπωρο θα είναι μια καλή στιγμή ενδεχομένω για το Κοινοβούλιο να διοργανώσει μια συζήτηση με τα εθνικά κοινοβούλια. Ενδεχομένω να υπάρχουν ήδη καλέ πρακτικέ. Για παράδειγμα, το Γερμανικό Κοινοβούλιο έχει ήδη οργανωθεί με ένα σωστό τρόπο. Ενδεχομένω λοιπόν θα μπορούσε να διοργανωθεί μια κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών για το θέμα αυτό. Δεν τίφερε θέμα για την ε, χαρακτήρα των προκλήσεων πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Χάζενκαμπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Από αλληλεγγύη με τους δερμηνείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μιλήσω στα Ολλανδικά. Αν πιστέψουμε τι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει, τα πράγματα πηγαίνουν όλα καλά και θα πετύχουμε του στόχους ε, της βιώσιμης αναπτυξικούς στόχους. Ωστόσο, στην πράξη τα πράγματα διαφέρουν. Η Ολλανδία, για παράδειγμα. Η Ολλανδία δεν θα πετύχει πολλού από του βιώσιμού αναπτυξιακούς στόχου. Έχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό όλο και πιο πολύ φτώχεια περιορισμένε ανανεώσιμε ενέργειε. Η γεωργία είναι οργανική και βιολογική σε περιορισμένο μόνο ποσοστό και τα του θερμοκηπίου είναι πολύ πιο υψηλά από ό,τι σε άλλες χώρες. Και δεν γίνονται οι απαραίτητε ενεργείες για να αντιμετωπίσει αυτή η κατάσταση. Θέλω σήμερα να ζητήσω προσοχή για τον ε, βιώσιμο αναπτυξιακό στόχο υπαριθμών 12 μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα κατανάλωσης και πραγωγής. Οι προσπάθειε για την κυκλική οικονομία αποτελεί, αποτελούν ένα καλό βήμα. Δεν αρκούν όμω. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατανάλωση κρέατος και ψαριού. Καταστροφική για τον πλανήτη, γιατί εκατομμύρια ζώα υποφέρουν περιτά και η βιομηχανική ε, κτηνοτροφία έχει ως αποτέλεσμα τη μόλυνση των θαλασσών, των εδαφών, τη μόλυνση των ε, ζώων και των ανθρώπων. 70% όλων των ε, πόσο υδάτων χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο για την κτηνοτροφία. Ένα κιλό, ένα κιλό κρέατος ε, κοστίζει 15.000 λίτρα νερό και η παραγωγή κρέατος είναι υπεύθυνη για 30% των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου και με τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται μπορούμε να ταΐσουμε 10 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο όμως αν έχουμε πιο πολύ ε, χορτοφαγική διατροφή. Βιώσιμη. Θα πρέπει να περάσουμε σε φυτικές ε, τροφές και θα πρέπει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκοπεύει να κάνει για να προωθήσει αυτή τη φυτοφαγική διατροφή. Πώς θα πετύχετε το στόχο υπαριθμών 12, αγαπητή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί με την κοινή αγροτική πολιτική και την καινούργια, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ απλά συνεχίζει τι παροχή κινήτρων στην κτηνοτροφία. Και η κτηνοτροφία έχει συνέπειε και για τον βιώσιμο αναπτυξιακό στόχο υπαριθμών 6. Γιατί είναι μέσα στα νετρικά το έδαφος μας και τα νερά μας και με φωσφορού χάλατα. Τι να πούμε δε και για τα ευρωπαϊκά προγράμματα αλίας. Ακόμα οδηγούν σε υπεραλίευση. Τι νομιμοποιούν κιόλας για παράδειγμα το σχέδιο για τη Βαλτική και για την Βόρεια Θάλασσα. Τι θα κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της αλίας και της ακτινοτροφίας και να μπορέσει να πετύχει κάποια στιγμή της βιώσιμης αναπτυξιακούς στόχους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακαβάνη, η συμπρόεδρος, να πάρει το λόγο. Έχει και αυτή μια ερώτηση να κάνει. Πρωτού κλείσουμε το γύρο αυτό των ερωτήσεων. Ευχαριστώ να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ακούσαμε διάφορους συναδέλφους ε, που μίλησαν. Και τι θα μας παρουσιάσει το 2019 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό θα να έχουμε λίγο μια σαφήνεια για το τι ακριβώς σκοπεύει να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο υψηλό βαθμό πολιτικό φόρουμ, γιατί Φανταζόμαστε ότι θα είναι κάποιε ιστορικές και κάποιες εξωτερικές πτυχές, ε, κάποιοι προσκεκλημένοι από το... Ο προσκεκλημένο από τη UMEPS νομίζω είπε ε, ότι για να παρακολουθήσουμε την πρόοδο που χρειάζονται ορόσημα. Έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορόσημα. Κάποια πολλά κράτη-μέλη έχουν κάνει τις εθνικές εθελούσιες ε, αναθεωρήσεις. Θα τις κοιτάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτές τις αναθεωρήσεις θα κάνει μια σύγκριση, κάποια ανάλυση για να δώσει και κάποια κίνητρα στα κράτη-μέλη. Ελπίζω να μην είναι απλά ένα σερτάρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μαζεύουμε ωραία ωραία όλες αυτές τις εκθέσεις. Να υπάρχει κάποια σύγκριση, γιατί αυτό που είπε η κυρία Ανελίτση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τη στιγμή που η πολυμέρεια είναι υπό επίθεση. Ο κόσμος περιμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ μας περιμένει να δώσουμε την κινητήριο δύναμη και την οθήση από την DG DEFCO. Θα πάρει το λόγο ο κ. Γκάσπερτ για να μας απαντήσει σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω πώς ε, σκοπεύετε να οργανωθείτε, ποιος ε, θα πάρει το λόγο ο Γενικός Γραμματέας θα συντονίσει την ε, δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο Ιούλιο, αλλά και ο κ. Φοντίνη ενδεχομένω να θέλει να πάρει το λόγο. Okay. Um, thank uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να πω δύο λόγια για το πώς ε, θα απαντήσουμε στην εξωτερική ε, πτυχή, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Συμφωνούμε όλοι ως προς αυτό. Όπως ξέρετε, οι βασικές ε, δράσεις για την εφαρμογή του εξωτερικού κομματιού ήταν ε, η δημιουργία μιας νέας συμφωνίας για την ε, ανάπτυξη. Ήταν το νέο πρόγραμμα, το νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη για να καλύψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη-μέλη. Και βεβαίως αυτό έχει συμφωνηθεί και από το Κοινοβούλιο. Τώρα λοιπόν έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να γραφτούν όλα αυτά, να μεταφραστούν σε πολιτική, να γίνουν ε, εκθέσεις, ε, πλαίσιο διεθνών συμφωνιών κτλ. Όπως αυτή που θα υπάρξει για τον έλεγχο. Και επίσης το πώς θα ε, υποβληθούν οι εκθέσεις για τον έλεγχο. Προβλέπεται λοιπόν αυτό στην συνένεση, μια έκθεση που θα αναφέρει πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της από κοινού υποστηρίζουν και βοηθούν τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες για την εφαρμογή του θεματολογίου και της Ευρωπαϊκής Συνένεσης. Θα το κάνουμε αυτό επί τη βάση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών που έχουμε. Θα υποβληθούν εκθέσεις για όλα τα στοιχεία, για την ε, ανάπτυξη την οικονομική, για τους BCDs, ε, για τα αποτελέσματα και βεβαίως θα ζητήσουμε και τη βοήθεια των κρατών μελών. Είναι κοινή αυτή η έκθεση με τα κράτη-μέλη και μπορούμε έτσι να έχουμε πιο ενοποιημένη προσέγγιση για τις ε, εθνικές εκθέσεις, τουλάχιστον για το καλοκαίρι, γιατί αφού θα κάνουμε από κοινού τις ε, αναφορές για την ε, εφαρμογή της συνένεσης, θα έχουμε και μια ιδέα γενικότερη του πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα των εκθέσεων και ελπίζω ότι έτσι θα μεταφερθούν και αυτά στις εθνικές ε, εκθέσεις των κρατών μελών. Ε, νομίζω λοιπόν ότι είναι κοινή η δράση αυτή και είναι και σημαντική για το εξωτερικό κομμάτι της ε, συνένεσης. Και επίσης επειδή υπήρχε ένα ερώτημα για την συνεκτικότητα των πολιτικών για την ανάπτυξη, προσπαθούμε να δουλέψουμε λίγο περισσότερα, και, λίγο καλύτερα μάλλον, και να προσαρμοστούμε ενσωματώνοντας πλήρως τη δουλειά που κάνουμε για το BCD στην ε, μέθοδο εργασίας της συνήθη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε την ε, διεπηρεσιακή ομάδα για, την, ε, για, την, το θεματολόγιο του 2030 και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποδοτικοί και θα χρησιμοποιήσουμε την ε, πολιτική, τη συνεκτική πολιτική ώστε να υπάρξει μια πιο ένα πιο ευρύ εγχείρημα για την βιώσιμη ανάπτυξη συνολικά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω ότι για μας το πολιτικό πλαίσιο για το 2019 την, στην Επιτροπή ε, Ανώτερων Αξιωματούχων. Το έγγραφο αυτό θα αντικατοπτρίζει τα πολιτικά πλαίσια λειτουργίας. Καθίσταται σαφές ότι ότι θα έχουμε μία ολοκληρωμένη παρουσίαση της εσωτερικής και εξωτερικής ε, διάστασης και αυτή τη στιγμή συζητάμε τη μορφή που θα γίνει μαζί με την ΕΙΕΔ επίσης. Δεν έχει αποφασιστεί η μορφή εσωτερικά. Άρα θα πρέπει να κάνετε υπομονή αλλά θα σας κρατήσουμε ενήμερους για τις προθέσεις Επιτροπής και της ΕΙΕΔ. Ως προς το έγγραφο περισύλλογής, μας ενδιαφέρει και το πλαίσιο εποπτείας για να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί. Ε, καθίσταται σαφές ότι δεν μπορούμε να εφευρίσκουμε νέους στόχους από το πουθενά. Οι στόχοι είναι πολιτικοί καθαρά. Αφορούν πολιτικές αποφάσεις, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Μετά από τις συζητήσεις για το κλίμα και το περιβάλλον. Άρα δεν πρόκειται για ένα γραφειοκρατικό εγχείρημα. Αφορά μια πολιτική συζήτηση και θα δούμε πώς μπορεί να γίνει κατά τον καλύτερο τρόπο. Και δεν θα ήθελα να υποβιβάσετε το ρόλο της Eurostat στην εποπτ και την πρόοδο προς τους ε, βιώσιμους στόχους. Η Eurostat ε, έχει αναλάβει την πραγματογνωμοσύνη αυτή συλλογή στατιστικών στοιχείων όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στα κράτη-μέλη και αυτή την ε, πραγματογνωμοσύνη, αυτή η πραγματογνωμοσύνη είναι ένα κοινό εγχείρημα ε, δεν θα πρέπει να γίνουν ε, εύκολες επικρίσεις ε, κατά της Eurostat. Όλη η εργασία της αφορά μία εντατική συνεργασία με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω ότι οι στόχοι έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Και γι' αυτό θα, θα τα πούμε στη Νέα Υόρκη ξανά. Είχαμε ε, συναντηθεί δύο χρόνια πριν. Το ζήτημα είναι οι τιμές αναφορές, αναφοράς για να δούμε κατά πόσο έχει επιτελεστεί η πρόοδος. Δηλαδή η Eurostat ε, δεν είναι να συλλέξει στατιστικές, αλλά τι θα κάνουμε εμείς όταν συλλέξουμε στατιστικές, πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε. Τι θα κάνουμε δηλαδή με τα λύματά μας. Στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο εξάγουμε πλαστικά στις φτωχές χώρες. Το θέμα αυτό είναι θέμα πολιτικής. Τι θα κάνουμε με τη συλλογή στοιχείων, τι θα κάνουμε τα στοιχεία που θα έχουν συλλεχθεί. Και με το έγγραφο περί συλλογής θα δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς ε, τη Νέα Υόρκη. Είπαμε θα το κάνουμε. Τέσσερα χρόνια μετά λοιπόν θα πρέπει να δείξουμε ότι κατέχουμε ηγετική θέση. Και αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό για τη διάσκεψη που θα γίνει. Νομίζω πρέπει να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ε, ομιλητές. Η κυρία Χάουταλα είχε απόλυτο δίκιο και όταν επανέλθει η αντιπροσωπεία από τη Νέα Υόρκη θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να ε, βάλουμε, να εντάξουμε ορισμένα στοιχεία στο έγγραφο περισυλλογής, γιατί αν το λάβουμε μετά τα Χριστούγεννα δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θα θέλαμε ο Επίτροπος ε, Τίμερμανς ε, να μας πει στην Ολομέλεια πώς, ε, τι πρόοδος έχει επιτελεστεί σε αυτό το έγγραφο περί συλλογής. Φαντάζομαι τον Οκτώβριο θα ξέρουμε τι θα γίνει για να μπορέσουμε και εμείς να έρθουμε σε επαφή με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πρόκειται για μια συλλογική πολιτική προσπάθεια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε το Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής. Ευχαριστούμε την Γενική Διάθεση ΔΕΦΚΟ, τον Γκασπάρ Φοντίνη. Και έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε τι προθεσμίες υπάρχουν και τι χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ τους πάνελιστ και την Επιτροπή. Δεν ξέρω κατά πόσο η κυρία Βαλέαν έχει κάτι να προσθέσει. Όχι, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι. Έχουμε πολλά θέματα προς αντιμετώπιση. Θα δούμε λοιπόν τι θα μας πείτε μετά τη Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε όλοι.